Με ακούτε τώρα? Με ακούτε όταν φοράτε τα ακουστικά σας. Λειτουργεί η διερμηνία. Το σύστημα επανήλθε. Πολύ ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι πρέπει καταρχάς να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 12 Σεπτεμβρίου, κάναμε μια τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη, γιατί στις 12 Σεπτεμβρίου είχαμε ένα αίτημα από την πολιτική ομάδα ECR. Επιβλήθη λοιπόν ένα αίτημα από την πολιτική αυτή ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 214 του κανονισμού, όσον αφορά τις συστάσεις των συντονιστών για το σημείο 4,4 από το έγγραφο των συντονιστών όσον αφορά την εξέταση μιας νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αντίρρηση, μπορούμε να εγκρίνουμε την τροποποιηθήσα ημερήσια διάταξη. Συμφωνούμε πολύ ωραία. Περνάμε στις ανακοινώσει. Έχουμε όλες τις γλώσσες διαθέσιμες, εκτός από μαλτέζικα, λετονικά και ιρλανδικά. Για τις γλώσσες αυτές δυστυχώς δεν έχουμε διερμηνία. Ας περάσουμε τώρα στο πρώτο νέο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Όπως σας είπα, υπευλήθη ένα αίτημα από το ECR. Σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουμε για την απόφαση των συντονιστών. Προκειμένου να εγκρίνουμε τι αποφάσεως των νηστών της συνεδρίασης της 5 η Σεπτεμβρίου. Ξέρετε ότι τότε αποφάσισαν να αποφανθούν για όλα τα αιτήματα υποβολής εκθέσεων πρωτοβουλία στη συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα τον Οκτώβριο. Ελήφθη λοιπόν μια απόφαση από του τονιστέ να αναβληθεί η λήψη απόφασης όσον αφορά τι εκθέσει πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν όλες οι εκθέσεις πρωτοβουλίες που έχουν προταθεί από τις διάφορες πολιτικές ομάδες θα αποτελέσουν αντικείμενο απόφαση στην επόμενη συνεδρία των τονιστών που θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο. Όμως το ECR αντετάχθη στην απόφαση αυτή. και πρότεινε να τροποποιηθεί η απόφαση αυτή των συντονιστών και κάναν ειδική μνήα στην απόφαση εκείνη που είχε να κάνει με το ένταλμα σύλληψης, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Να δώσω λοιπόν καταρχάς το λόγο στον εκπρόσωπο του ECR που θέλει να μιλήσει για το ζήτημα αυτό και μετά θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα λόγια σας και να τονίσω προς όλα τα μέλη της Επιτροπής που δεν ήταν στις Βρυξέλλες ε, να εξηγήσω το λόγο για το οποίο ζητήσαμε αυτή τη διαδικασία. Η πρότασή μας είναι μετά από μια έκθεση νομο, ιδίας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση και βελτίωση του συστήματος του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που δύο φορές ε, αμφισβητήθηκε από τους συντονιστές 24 Ιουλίου και 5 Σεπτεμβρίου και εμείς θεωρούμε ουσιαστικό βασικό κομμάτι του ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι να εμποδίσει χιλιάδες ε, ε, παράνομοι να αποφεύγουν την καταδίκη από κυρία Χακράτη περνώντας από τα σύνορα και εκμεταλλευόμενοι τον ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης σεβόμαστε, μιας, πρέπει να σεβόμαστε μια σειρά αποφάσεων και ε, μπορούμε κάλλιστα να προχωρήσουμε τώρα. Αυτό αφορά σε περίπτωση που υπερψηφιστεί το αίτημά μας θα πρέπει να εννοηθεί ότι υπάρχει εντολή της Επιτροπής να προχωρήσει στην βελτίωση αυτού του κειμένου. Ακούσατε την άποψη του εκπροσώπου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών πρόκειται για απόφαση του, των συντονιστών στις 12 Σεπτεμβρίου να αποφασίσουμε για τις διάφορες προτάσεις ίδιας πρωτοβουλίας μόνο στην επόμενη συνάντηση τον Οκτώβριο. Δεν επηρεάζει δηλαδή το θέμα, δεν επηρεάζει την ουσία, επηρεάζει μόνο τον τρόπο που θα προχωρήσουμε, το διαδικαστικό. Προτείνω λοιπόν την εξής διαδικασία. Πρώτον, ψηφίζουμε με την ακόλουθη διαδικασία. Αν είστε υπέρ των αποφάσεων των συντονιστών που λήφθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του συγκεκριμένου αιτήματο των συντηρητικών μαζί με τα υπόλοιπα θέματα ίδιας πρωτοβουλία να αποφασιστούν στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών 8 Οκτωβρίου ή ψηφίστε υπέρ της απόφασης των συντονιστών. Ναι, συν με την ηλεκτρονική σας ε, ε, κάρτα. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Να έχετε μαζί σας την κάρτα σας. Αλλιώς στείλτε κάποιον να σας τις φέρουν. Αν υποστηρίζετε το αίτημα του ECR να διαχωριστεί η συγκεκριμένη έκθεση δύο πρωτοβουλίε από το υπόλοιπο πακέτο που πρέπει να αποφασιστεί στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών, ψηφίζεται μείον, πλην, αρνητικά. Συν αν είστε υπέρ της θέσης των συντονιστών, πλην αν είστε υπέρ της θέσης του ECR. Ήμπο, για να πόσχετε βέβαια. Αυτή είναι η διαδικασία. για να το διευκρινίσω. Αν κερδίσει το πλήν, θα υπάρξει απόφαση ως προς την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Αν όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει έκθεση ιδίε πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, γιατί αυτό θα το αποφασίσουν οι συντονιστέ τον Οκτώβριο με το υπόλοιπο πακέτο. Έγινε σαφή. Υπέρ τη θέση των συντονιστών συν κατά πλην. Open the vote. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπάρχει ένας επιπλέον από τους σοσιαλιστές από ό,τι φαίνεται. Ένας λιγότερος σοσιαλιστής, παρακαλώ. Ακόμα ένας. Πέρας ψηφοφορίας. 50 against 7, so it means that... 50 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνονται λοιπόν οι θέσει των συντονιστών. Όλες οι αποφάσεις για τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας θα γίνουν τον Οκτώβριο. Διευκρινίζω εκ νέου ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, αλλά ότι αυτό θα αποφασιστεί τον Οκτώβριο. Προχωρούμε. Στην προηγούμενη μερίσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων με τον αγαπητό επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Υπεύθυνο για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών και ηθαγένειας. Τον καλωσορίζουμε με χαρά στην Επιτροπή ξανά είχαμε ανταλλαγή απόψε με την Επίτροπο για, την δικαι... για τα θέματα δικαιοσύνη στην κυρία Γιούμποροβα, τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντ, τον Τζούλιαν Κίνγκ για τα θέματα ασφάλεια. και ακούμε το, θα ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο. Φεύγει Σιγά σιγά τον ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που έκανε τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο συζητήσεων, ερωτήσεων από τους συντονιστές, δύο λεπτά και κατόπιν θα δούμε ποια μέλη θέλουν να λάβουν το λόγο. Όταν μετρήσουμε τα ονόματα θα δώσουμε το χρόνο ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο περισσότερους γίνεται να μιλήσουν. Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω να παρουσιάσετε, καλωσορίζω να παρουσιάσετε τις τελευταίες απόψεις για το χαρτοφυλάκιό σας. Και σας καλωσορίζω εκ νέου στην Επιτροπή ΛΥΜΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι η πρώτη φορά κατά τα πέντε τελευταία χρόνια που απευθύνομαι σε αυτή την Επιτροπή με τη νέα της σύνθεση μετά τις ευρωεκλογέ και είναι και η τελευταία φορά επίσης. Αλλά θεωρώ ότι με την σημερινή ευκαιρία ε, θα, θα πρέπει να σας χαιρετήσω και να σας πω και αντίο. Η συζήτησή μας σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να αναγνωρίσουμε πόσο μακριά έχουμε προχωρήσει κατά τα πέντε τελευταία χρόνια και επίσης να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, προκλήσεις για σας. Είμαι ευτυχής που Είδα ότι αναλάβατε κύριε Πρόεδρε εσείς τα καθήκοντά σας άλλη μια φορά η Προεδρία ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Νομίζω ότι οι δεσμεύσει σας, η πείρα σας, το παρελθόν σας αλλά επίσης ε, και τα βιώματα, τα πολιτικά που έχετε από το παρελθόν θα είναι πολύτιμα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω ε, στον Μωράς τον φίλο μου, τον πρώην ε, πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, για την εξαίρετη συνεργασία και δέσμευση για αποτελέσματα για φιλόδοξα ε, σχέδια κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Κοινοβουλίου. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία Είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει ως το τέλος της θητείας μου ως Επιτρόπου και ακόμη πιο σημαντικό είμαι βέβαιος ότι η φιλία που είχα την ευκαιρία να έχουμε πολλούς από εσά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών θα συνεχιστεί για πολύ περισσότερο χρόνο. Ε, χαίρομαι που ε, ανήκετε σε αυτήν την Επιτροπή, διότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει ζωτικό ρόλο να παίξει για την πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική μετανάστευσης και ασφάλειας για τις προκλήσεις αυτές που θα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο με κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Πάρα πολλά έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών με την υποστήριξη και την βοήθεια του Κοινοβουλίου και κυρίως της δυναμικής σας Επιτροπής. Είμαι ευγνώμων ε, στους συναδέλφους σας. Θυμάμαι όταν αρχίσαμε μαζί την εργασία, τη συνεργασία με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ε, έπρεπε όταν ε, ορίστηκα επίτροπος σε σε πέντε μήνες έπρεπε τα βασικά θέματα του χαρτοφυλακίου μου, τη μετανάστευση, την ηθαγένεια και εσωτερικής υποθέσεις να είναι προτεραιότητα της Επιτροπής. Ε, δεν ξέραμε και στα κράτη-μέλη πώς να βοηθήσουμε την κατάσταση, αλλά με τη συνεργασία μπορούμε να πούμε σήμερα ότι έχουμε πράξει πολλά αλλά υπάρχουν και πολλά που πρέπει ακόμη να γίνουν στο μέλλον από τις 2015 είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις στον ε, τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Με εμονή, με επιμονή κατορθώσαμε σε λίγα χρόνια να έχουμε όλα στα απαραίτητα εργαλεία και να έχουμε μια εύρωστη πολιτική για το μέλλον. Και η εργασία αυτή πρέπει να συνεχιστεί, διότι και τα δύο θέματα θα θα υπάρχουν ακόμα έχουμε προτείνει μέτρα αμέσως για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση και απάντηση στην κρίση ε, και λύσεις για καλύτερη αντιμετώπιση εσωτερική και εξωτερική της μετανάστευσης ε, για να σώσουμε ζωές. Πάνω από 700.000 ζωές σώθηκαν από το 2015 στην Μεσόγειο, υποστηρίζοντας τα κράτη-μέλη με μεγάλη πίεση ε, για να λάβουν, να υποδεχθούν ε, τους μετανάστες, δίνοντας υποστήριξη οικονομική και τεχνική επιτόπου ούτως ώστε να γίνει η επανεγκατάσταση μια πραγματικότητα. Πάνω από 34.000 άτομα έχουν επαναγκατασταθεί από την, στην Ελλάδα και Ιταλία και στην Ευρώπη από, ε, από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016. Ε, μείωση των κινήτρων για την παράνομη μετανάστευση καταπολέμηση των διακινητών παράνομων μεταναστών ε, και βοηθώντας ε, τις χώρες προέλευσης ε, και διέλευσης από κάθε άποψη. Σήμερα οι αριθμοί των παράνομων αφήξεων είναι κάτω από την εποχή της κρίσης. Η ενίσχυση και εξυγχρονισμός ε, της διαχείρισης ε, των συνόρων, ούτω ώστε να διευκολύνουμε αυτούς που έρχονται καλή την πίστη. Θέλουμε να έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου για να ενισχύσουμε την πολιτική επιστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να βοηθήσουμε για την νόμιμη μετανάστευση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ένα σημαντικό σημείο της πολιτικής μας ήταν να ενισχύσουμε ε, τα μέσα, τα νομικά για τα άτομα που χρήζουν ε, διεθνούς προστασίες και για αυτούς που έχουν οικονομικές ανάγκες. Αυτό είναι καλό για να μπορέσουμε να αποθαρρύνουμε τους παράνομους δρόμους και να έχουμε ένα business model και να βοηθούμε να προσελκύσουμε τα άτομα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες που βοηθούν την οικονομία. Είναι λυπηρό ε, ότι δεν ήταν δυνατόν να συμφωνήσουμε για μια ε, καλύτερη μπλε κάρτα του Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και τους καλούς εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές. Αλλά η ανάγκη ε, για μια, ένα ελκυστικό ε, σχέδιο για τους πιο ταλεντούχους για να βοηθήσουμε την αντιγωνιστικότητα της οικονομίας μας και να διευκολύνουμε την μετανάστευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να παραμείνει. Νομίζω ότι το νέο κοινοβούλιο θα κρατήσει το ίδιο επίπεδο φιλοδοξία σχετικά με το θέμα αυτό. Ένα κεντρικό μέρος της πολιτικής μας υπήρξαν και οι συνέργειες μας με χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε στην ανάγκη να ενισχύσουμε συμπράξεις μακροπρόθεσμες με χώρες προέλευσης και διέλευσης για να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες, τις ε, αιτίες ε, των, ε, της μετανάστευσης για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες και να αντιμετωπίσουμε τη λαθρέα διακίνηση μεταναστών για να διευκολύνουμε την ένταξη, για να προσαγάγουμε στην δικαιοσύνη τους διακινητές και να διευκολύνουμε τις, τα νομικά μέσα. Πάρα πολλά προγράμματα πιλωτικά ε, τώρα εκπονούνται και νομίζω ότι μερικά κράτη-μέλη έχουν ε, συμμετάσχει. Η δήλωση και της Τουρκίας ε, και η συμφωνία μείωσε τις ροές μεταναστών κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα αυτό με την Τουρκία αποτελεί κεντρικό σημείο της συνεργασίας μας ε, για την διευκόλυνση των συνθήκων ζωής και για τις ε, συνθήκες στην Τουρκία. Παραδείγματο χάρη έχουμε δώσει πρόσβαση στην εκπαίδευση σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών της Συρίας και εκατομμύρια έχουν λάβει βοήθεια για τις καθημερινές τους ανάγκες. Η υποστήριξή μας βοήθησε στην οικοδόμηση εγκαταστάσεων υποδοχής και υγειονομικών εγκαταστάσεων. Σε σχέση με τις θεωρήσεις που νομίζω ότι ήταν το αγαπημένο σας θέμα κύριε Πρόεδρε, κατορθώσαμε να βρούμε μια συμφωνία για την αναθεώρηση των θεωρήσεων που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου. Η νέα πολιτική των θεωρήσεων θα ενδυναμώσει ε, την, ε, την, ε, τα σύνορα και τις, θα μειώσει τους κινδύνους και θα βοηθήσει όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται καλή την πίστη. Παραδείγματο χα, την Γεωργία, από την Ουκρανία τώρα μπορούν να έρθουν στην ε, περιοχή Σέγγεν χωρίς θεωρήσεις. Αυτό είναι ένα βήμα για να ενισχύσουμε τις δεσμούς με τις χώρες αυτέ. Ταυτόχρονα η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων. Και τώρα θα ήθελα να στραφώ ε, σε ένα από τα σφακέλους τους πιο σημαντικούς που θα αποτελέσει πραγματική αλληλεγγύη για την μετανάστευση, η εγκατάσταση μια, ενός κοινού ε, συστήματος ευρωπαϊκού ασύλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της προηγούμενης ε, κοινοβουλευτικής περίοδου γιατί ε, ενέκριναν ε, συγκεκριμένη θέση και για τις επτά νομοθετικές προτάσεις και γιατί δείξαν ότι πραγματικά ήθελαν να συνεργαστούν με το Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθούν όλες αυτές οι προτάσεις. Επιγόντως χρειάζεται να αναθεωρηθεί η πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνη προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό κοινό σύστημα ασύλου. Γιατί αυτό λειτουργεί προ το συμφέρον όλων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τις α, διάφορες περιπτώσεις μόνο κατά περίπτωση και δεν μπορούμε να δείχνουμε μόνο την αλληλεγγύη κάθε φορά που προσεγγίζει τις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σκάφος. Βασίζομαι λοιπόν σε εσά προκειμένου να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προκειμένου να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για βιώσιμες λύσεις, ιδίως όσον αφορά τις επόμενες βαθικέ προτάσεις για τη μετανάστευση και το άσυλο, όπως το ανακοίνωσε η νεοκλεγήσα πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος μας είναι να έχουμε έναν μηχανισμό βιώσιμο, ένα μηχανισμό λιλεγγύης που θα αποτελεί τμήμα ενός μόνιμου μηχανισμού λιλεγγύης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κοινού συστήματος ασύλου και συγκεκριμένα στα πλαίσια του νέου κανονισμού Δουβλίνου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε εκ νέου τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να επαναγκαταστούν κατά εθελούσια βάση με χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρουμε να εγκρίνουμε εν τέλει ένα νέο κανονισμό Δουβλίνου. Αρκετά άλλα πάντα τα ίδια τελικά κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία ανταποκρίθηκαν θετικά στην έκκληση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία προχώρησαν σε δράσεις μετεγκατάστασης μετά από αποβιβάσεις που γίναν το 2018 και το 2019. Μετά τα συμβάντα απόβασης που είχαμε στην Ιταλία τον Ιούνιο του 2018 και το Σεπτέμβριο, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2019 εν συνεχεία, χίλια άτομα έχουν μεταφερθεί σε άλλα κράτη-μέλη και στην Νορβηγία, σύμφωνα με τις εθελούσιες δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι συγκεκριμένε αυτές χώρες τις οποίες ανέφερα. 760 τώρα άτομα μεταφέρθηκαν από την Μάλτα και 240 από την Ιταλία έως 855 ε, άτομα για, 800, για έως 855 άτομα εκκρεμούν ακόμα οι αιτήσει ε, κατάσταση και επί του παρόντος εξελίσσονται συζητήσεις προκειμένου να καταφέρουμε να ευθυγραμμίσουμε τα αιτήματα αυτά μέσω κάποιων προσωρινών διευθετήσεων καταλήγοντας όμως σε μια πιο συντονισμένη ανταπόκριση όσον αφορά τις ε, αποβάσεις αυτές. Και αυτό είναι ο στόχος τη συνάντηση που θα λάβει χώρο, την, την χώρα την επόμενη Δευτέρα στη Μάλτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδιάκοπα εργαζόταν τους τελευταίους μήνες προκειμένου να καταλήξει σε αυτές τις προσωρινές διευθετήσεις. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές μέχρι το τελευταίο λεπτό της θητείας μας, προκειμένου να εγκαθιδρυθούν αυτές οι λύσεις. Παρ' όλα αυτά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στη θέση της ότι θα πρέπει να έχουμε μία μόνιμη και διαρθρωμένη λύση η οποία να είναι αναπόσπαστο τμήμα του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το συντομότερο δυνατό. Επίσης, ένα βασικό συστατικό μία ισορροπημένης και αξιόπιστης πολιτικής ε, ασύλου είναι αυτή η οποία θα προβλέπει και ένα σύστημα επιστροφής για όσους δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς κάνουμε κάθε το δυνατό για να επεμβαίνουμε το συντομότερο δυνατό για να αποτρέψουμε την παράτυπη μετανάστευση και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια τη μετανάστευση αυτή. Στην περίπτωση όμω των ατόμων εκείνων, εκείνων που διαμένουν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άτομα αυτά θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να επιστρέφονται στι χώρε προέλευση σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθώντας βέβαια πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αυτών. Προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε λοιπόν αποτελεσματικού μηχανισμού για τέτοιε επιστροφέ, καλώ την Επιτροπή σα να ξεκινήσει εκ νέου τι εργασίε τη όσον αφορά την αναθεώρηση τη οδηγία επιστροφών το συντομότερο δυνατό. Ε, μια ακόμα προπόθεση για να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που να λειτουργεί είναι ένα χώρο Σέγγεν, ο οποίο να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ξέρετε ότι ο χώρο Σέγγεν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρώπη σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιστρέψει στην παρελθούσα κατάσταση. Δεν μπορούμε να ζούμε ως Ευρώπη με κλειστά σύνορα. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό και θα πρέπει να γνωρίσουμε και ποια είναι η στάση ορισμένων κυβερνήσεων και όχι κρατών μελών, η στάση ορισμένων κυβερνήσεων και μένω σε αυτό. Εξαιτία τη στάση ορισμένων κυβερνήσεων κινδυνεύει ο χώρο Σέγγεν. Εμεί καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προασπίσουμε, να προστατεύσουμε τον χώρο Σέγγεν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν χώρο Σέγγεν ο οποίο να λειτουργεί πλήρω όπω το παρελθόν. Και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ξεκάθαρου κανόνε για τα κράτη-μέλη όσον αφορά του ελέγχου στα εσωτερικά του σύνορα που θα πρέπει να βασίζονται σε ένα καθεστώ εμπιστοσύνη όπω είπαμε πριν από λίγο. Θα πρέπει όμω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή και η κυρία Φαγιόν είμαι σίγουρος ότι ε, παραμένει και αυτή προσιλωμένη στο στόχο αυτό. Η προστασία τώρα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λειτουργία του χώρου Σέγγεν θα ενισχυθούν από το νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με μόνιμες δυνάμεις 10.000 και με πραγματικές αρμοδιότητες για να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη. Προσβλέπω λοιπόν στην γρήγορη και επίσημη έγκριση του σχετικού κανονισμού, προκειμένου η εργασία αυτή που εγκρίθηκε από τους νομοθέτες να αρχίσει να τίθεται σε ισχύ ευθύ αμέσω, προκειμένου πραγματικά να ανταποκριθούμε στη φιλοδοξία που έχει θέσει το νομοθετικό αυτό κείμενο. Τα εξωτερικά μας σύνορα αποτελούν πραγματικά το σύνδεσμο ανάμεσα στην όλη εργασία που έχουμε κάνει όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Χάρη στα επιτεύγματα της προηγούμενης νομοθετικής θητείας του προηγούμενου Κοινοβουλίου, όλα τα άτομα τα οποία διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάνε από προηγμένα συστήματα ελέγχου, όπως το σύστημα Schengen, το Ευρωπαϊκό Σύστημα για τα Ταξίδια και την Αδειοδότηση, καθώς επίσης και το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου. Ξέρετε ότι τα συστήματα αυτά ελέγχου δεν υφίστανται, δεν υφίσταντο στο παρελθόν. Επομένως, τα σύνορά μας τώρα τη χάνουν καλύτερης διακυβέρνησης, καλύτερης προστασίας, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το στόχο αυτό. Το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τα συστήματα αυτά. Η διαλειτουργικότητα λοιπόν, η οποία θα διασυνδέει όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα, αποτελεί το τελευταίο επίτευγμα το οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα προκειμένου να μην λειτουργούμε με τρόπο κατακαιρματισμένο, να είμαστε σε συνεχή επαφή μεταξύ ημών και να υποστηρίξουμε καταλήλω τα σημεία άφηξη, όπω και πράγμα του λιμένε. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται με τα κράτη-μέλη μέσω του συστήματο EU-LISA, προκειμένου να έχουμε μια γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων αυτών συστημάτων που θα πρέπει όμως και να συνομιλούν μεταξύ τους. Θα πρέπει γι' αυτόν τον λόγο να καταλήξουμε νωρίς το 2020 σε μια συμφωνία όσον αφορά τον νέο Ευρωπαϊκό Κώδικα Θεωρήσεων, προκειμένου να μπορεί και αυτός να συντονιστεί με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας που έχουν τα υπόλοιπα συστήματα. Δεν θα παριθμίσω αυτή τη στιγμή όλε τι νομοθεσίες που έχουμε εγκρίνει στον τομέα της ασφάλειας. Όπως είχατε υποδεχθεί τον Επίτροπο Κίνγκ στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής σας, και καθότι γνωρίζω ότι σας έκανε μια παρουσίαση για τα συστήματα αυτά ασφαλείας, το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει να επιτεχύνουμε τον προγράμμα δυνατό την έγκριση όσον αφορά την έγκριση του νομοθετικού φακέλου για το περιεχόμενο τρομοκρατικής φύσης το επιγραμμικό. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι διαφορετικές επιγραμμικές πλατφόρμες τις οποίες ελέγχουμε λειτουργούν σωστά. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε ένα σφαιρικό σύστημα το οποίο θα μπορεί πραγματικά να ελέγχει όλες αυτές τις πλατφόρμες όπως το Facebook και πολλές άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα πολύ πιο προστατευμένο πλαίσιο με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι τρομοκράτες να φεύγουν από μια πλατφόρμα και να εμφανίζονται σε μια άλλη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες μικρές πλατφόρμες οι οποίες δεν έχουν δηλώσει ακόμα την ενεργή συμμετοχή τους στο σύστημα αυτό. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα αυτό πείθοντα όλες οι πλατφόρμες να ενταχθούν στο σύστημα αυτό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το σημαντικό του αυτό ζήτημα. Κάποιες τελευταίες εξελίξεις, όπως ε, οι επιθέσεις που είχαμε στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας, έχουν καταδείξει την ανάγκη για ένα νομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταφέρουμε να επιταχύνουμε την νομοθετική μας ανταπόκριση όσον αφορά την επιγραμμική κατάχρηση του διαδικτυακού χώρου από τους τρομοκράτες. Και πραγματικά θα προσβλέπω στη θετική συνεργασία που θα έχουμε με τον κύριο Γιάκη για το ζήτημα αυτό. Επίσης, είναι σημαντική η περαιτέρω συζήτηση για την τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, κάτι το οποίο, με το οποίο ασχολείται η κυρία Ζίπελ. Περίπου οι μισές ε, ποινικέ έρευνες απαιτούν διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, άρα χρειαζόμαστε τα απαραίτητα μέσα για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Τελευταίο, σημαντικό, χρηματοδότηση. Η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση του μακροχρόνιου, της μακροχρόνιας χρηματοδότησης από το 2021 στο 2027 για το θέμα τα μετανάστευση και ασύλου, την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την ασφάλεια. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της με επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης. Ελπίζω ότι το νέο κοινοβούλιο θα κρατήσει ζωντανό το επίπεδο αυτό φιλοδοξίας. Συνάδελφοι, αυτές είναι κάποιες από τις συγκεκριμένες δράσεις και κάποια από τα συγκεκριμένα επιτεύγματα των προηγουμένων ετών που αποτελούν θεμέλιο για περαιτέρω δράση που ακόμα χρειάζεται. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας σε αυτό στόχος μας πρέπει να είναι να ολοκληρώσουμε και να συμπληρώσουμε την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο θέμα της μετανάστευσης και στο θέμα της ασφάλειας. Είναι καιρό τώρα να δώσουμε το, ε, τις αρμοδιότητες στην νέα Επίτροπη. την κυρία Γιώχανσεν. Πολύ δουλειά χρειάζεται να γίνει ακόμα. Το έργο της Επιτροπής θα συνεχιστεί με την ίδια ταχύτητα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από πλευράς μας κάναμε ό,τι μπορούμε, ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες, ιδίως στο ξεκίνημα της περίοδου. Θα, θα θυμούνται τις σκληρές στιγμές που περάσαμε ε, κάποιοι παλιοί από εσά στο ξεκίνημα του 2015 και στο ξεκίνημα του 2016. Δεν τα θυμάστε αυτά. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι όλοι, γιατί αφήσαμε πίσω μια κληρονομιά και η μετανάστευση και τα θέματα ασφάλειας θεωρούνταν στο παρελθόν ζητήματα κατά βάση εθνικών αρμοδιοτήτων. Σύντομα έγινε κατανοητό ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα με μια παγκόσμια διάσταση. Γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε στην αρχή ότι εδώ πρέπει να σκεφτόμαστε, να δρούμε και να ελοποιούμε αυτά που κάνουμε με ευρωπαϊκό τρόπο προς το όνομα όλων των Ευρωπαίων πολιτών όλων των ευρωπαϊκών εθνών. Πετύχαμε αλλαγή, μεγάλη αλλαγή αυτής της νοοτροπίας, δουλεύοντας με βασικά ευρωπαϊκές λύσεις, ενισχύοντας κάτι που αυτό δεν ήταν εύκολο, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, ενισχύοντας την ασφάλεια μεταξύ θεσμικών οργάνων και κρατών μελών. Επαναλαμβάνω ότι στον τομέα της ασφάλειας πέρασαμε δύσκολες στιγμές κατά την περίοδο 2015-2016 και αναπτύσσουμε τα κράτη-μέλη για την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών, για τη σύνδεση όλων των σημείων. Τα αποτελέσματα ωστόσο δείχνουν ότι πετύχαμε κάποια πράγματα. Κάναμε έναν πιο συνεκτικό τρόπο στην προσέγγιση μας ως προς την εξωτερική διάσταση της πολιτικής μας. Παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν όπως είπα. Θέλω εκ νέου να ευχαριστήσω όλους σας για τη συνεργασία στην υλοποίηση αυτών των συγκεκριμένων απαντήσεων στα ζητήματα πολιτικής βάσει των ευρωπαϊκών μας αξιών. Προσβλέπω στο να συνεργαστούμε μέχρι το τέλος της θητείας μου για να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε εκρεμή νομοθετικά κύματα στο μέτρο του δυνατού και είμαι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ερώτηση έχετε σήμερα αλλά και για τον υπόλοιπο μήνα της θητείας μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Τα τελευταία πέντε χρόνια εκφράσατε πραγματικά την σημασία του χαρτοφυλακίου σας σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς σας που είναι αρμοδιότητα και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, μετανάστευση, άσυλο και ανοίξατε δρόμο για συζητήσεις σίγουρα και είχαμε συζητήσει όλες τις συναντήσεις μετά από κάθε παρουσίασή σας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα έχουμε και τώρα συζητήσεις ξεκινούμε με τους συντονιστές δύο λεπτά ο καθένας γιατί υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος άλλων μελών που θέλουν το λόγο δύο λεπτά οι συντονιστές η κυρία Μετσόλα πρώτη Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο για τη σκληρή δουλειά που έκανε αλλά και το χιούμορ που κράτησε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές και την συνεχή βούλη συνεργασίας σας τα τελευταία χρόνια. Εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι έχετε κάνει, το έχουν πει και πολλοί συνάδελφοι στην αίθουσα, ανεξάρτητα από πολιτική ομάδα. Αυτά που μας είπατε είναι μια πλήρης ε, λεπτομεριακή εξήγηση του ιστορικού του έργου σας, αλλά όπως είπατε και εσείς έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να γίνει μπροστά και θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία για, που πρέπει να προχωρήσουμε όχι μόνο μέχρι το τέλος της, φοιτή, ε, της φοιτίας σας, αλλά και κατά την επόμενη πενταετία. Μπορούμε να πούμε ότι χάρη εμπολής και στη δική σας δουλειά θεσπίσαμε πράγματα που ήταν αδιανόητα πριν από λίγα χρόνια για την ε, διάσωση ανθρώπων, τη μείωση του τράφικινγκ και της διακίνησης ανθρώπων, την ταχύτητα στην επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πρόκρισης, ωστόσο η κατάσταση αυτό το καλοκαίρι στη Μεσόγειο συνεχίζει να είναι ανησυχητική. Υπάρχει κόσμος που χάνει τη πολίτες που χάνουν τη ζωή τους, υπάρχουν κράτη που εμποδίζουν την αποβίβαση ευάλωτων ατόμων. Είδαμε ε, πλοία με μπλοκαρισμένα στη θάλασσα, ανθρώπους να πηδούν στη θάλασσα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόσωπο της Ευρώπης που θέλουμε να δείχνουμε προς τον κόσμο. Τι θα κάνουμε, πώς θα έχουμε μια πιο αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, πώς θα έχουμε καλύτερη απόδοση στις επιστροφές, πώς θα έχουμε ε, καλύτερη λειτουργία των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την ε, μετεγκατάσταση των ετούντων. Έχουμε δει ότι το Δουβλίνο έχει μπλοκάρει από κάποια κράτη-μέλη. Μιλάτε λοιπόν για συστήματα αναδιανομής, για πιο αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι συμβουλεύετε την Επιτροπή αλλά και όλους μας. Παρακολουθώ τις συζητήσεις και στα άλλα θεσμικά όργανα που υπάρχει το μπλοκάρισμα στα βασικά εργαλεία. Ο κύριος Μωράης για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ε, βεβαίως είναι σύμπτωση που, ε, που βρίσκομαι εδώ, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, ε, αλλά χαίρομαι που είμαι εδώ για να εκφράσω την εκτίμησή μου στον Επίτροπο και ε, επικροτώ τα όσα είπε η κυρία Μετσόλα. Από την ομάδα μου εκφράζω την εκτίμησή μας, την προσωπική μου εκτίμηση για τα πέντε τελευταία χρόνια για το θέμα ασύλου. Έχουμε την συμφωνία με την ε, Τουρκία, έχουμε τα hot spots στην Ιταλία, έχουμε την κρίση όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά επίσης και στην ε, υπηρετική χώρα, ε, στην Γερμανία. Όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Αναφερθήκατε στις αλλαγές, αλλά αναφερθήκατε και σε εμά. Νομίζω ότι υπήρξε μια, δεν υπήρξε πάντα λογοδοσία προς αυτήν την Επιτροπή και υπήρξαν διάφορες ε, διαμάχες όπως θα συμφωνήσει και ο Πρόεδρος. Και θα ήθελα να εξφράσω για αυτήν την, τη σκληρή δουλειά που έκανε ο Επίτροπος και για τις αναφορές του. Η ερώτηση από την ομάδα μου είναι περίπου παρόμοια με της κυρίας Μετσόλα, ενώ ασχολείστε με την διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, το Σέγγεν. Έχουμε λοιπόν αυτήν την ε, κληρονομιά που αφήνεται σχετικά με το άσυλο και την μετανάστευση. Ε, το θέμα είναι ε, για τη νέα Επιτροπή και την, το τι αφήνεται πίσω για την νομική, τα νομικά θέματα της μετανάστευσης, αλλά πώς το Συμβούλιο θα μπορέσει να κινηθεί με ό,τι προβλέπεται στις συνθήκες και όλες τις προτάσεις που τις, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες για να υποστηρίξουμε την υπηρεσία ασύλου και αλλά βεβαίως έχουμε προσωρινά μέτρα, θα είναι πάντοτε προσωρινά τα μέτρα. Ε, τι θα γίνει με το μέλλον σύμφωνα με τα όσα έχουμε κληρονομήσει. Κυρία Review Europe. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Αβραμόπουλο. Είχα πάρα πολλά χρόνια την ευκαιρία να εργαστώ μαζί σας ακόμα και στην προηγούμενη θέση σας και σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για την μετανάστευση, διότι λέχθηκαν πολλά από τους συναδέλφους. Οι περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα ή αυτοί που αντιπροσωπεύουν το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν βρίσκονται όλοι στο ίδιο μήκο κύματο. Θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι παρά το γεγονός ότι 700.000 άτομα διασώθηκαν στην Μεσόγειο, χιλιάδες πέθαναν επίσης στην Μεσόγειο. Πάρα πολλοί χιλιάδες έχουν ε, μείνει στις, ε, στις, στα ελληνικά νησιά, σε, σε καταβλισμούς, στη Λιβύη, οι οποίοι δεν ξέρω μπορούν να θεωρούνται καταβλισμοί. Έχουμε λοιπόν αποτυχίες. Ξέρουμε ότι το θέμα το πρέπει ε, να λυθεί από το Συμβούλιο, διότι απορρίπτει κάθε απόφαση, αρνείται να λάβει κάθε απόφαση. Ε, και αυτό είναι μια αποτυχία. Η Επιτροπή έχει εξετάσει γιατί δεν το προσωρινός μηχανισμός προστασίας δεν έχει ε, ε, αρχίσει και γιατί αυτός ο μηχανισμός δεν θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ. Και ένα άλλο θέμα ένα θέμα που είναι και της ευθύνη σας. Έχουμε το πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις θεωρήσεις έχουμε ανάμεσα ότι θα χρειαζόταν ελεύθερα ταξίδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό λέχθηκε από το 2016. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα από την Ανατολική Ευρώπη που αποκλείονται από αυτήν την άδεια ε, και θα έπρεπε να γίνει μια αναφορά σχετικά με το θέμα αυτό. Τι έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό και αναφέρετε ε, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά ε, στοιχεία και όλα αυτά τα μέσα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων μας. Ε, ας δούμε την Δανία όπου χρειάστηκε να αναθεωρώσουν 10.000 αποφάσεις δικαστικές άτομα που αδίκως καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν επειδή ε, βασίστηκαν ε, σε αυτά τα δεδομένα. Δεν θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίδετε έστω και μια ευκαιρία να ανταλλάξω λίγο κάποιες απόψεις μαζί σας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε πραγματικά από κοινού με τα κράτη-μέλη να βρούμε λύσεις για τις προκλήσεις που υπάρχουν κυρίως στο ζήτημα της έρευνας και διάσωση. Είπατε για το 2015 όταν χιλιάδες Σύριοι ψάχνανε διεθνή προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά αφήσαμε την τουρκική κυβέρνηση να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Εσείς ασκήσατε τότε πίεση στην ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα προκειμένου να μπορούν να επιστρέψουν εκεί οι πρόσφυγες. Ο κύριο Ερντογάν όμως είπε ότι θα δημιουργήσει τώρα συγκεκριμένε ζώνες προστασίας στα βόρεια της Συρίας και λέει ότι ενδεχομένω θέλει να αποστείλει προ τα πίσω και τον εκατομμύριο Σύριου. Μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χέγγια αυτή τη στιγμή που ισχύουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο σιωπεί και θα μπορούσε να μα εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ακόλουθο. Αν θεωρεί την Τουρκία ω ασφαλή τρίτη χώρα, τότε μήπως θα έπρεπε να έχουμε μια πιο πρόσφατη έκθεση προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, γιατί η τελευταία τέτοια έκθεση είναι από το Μάρτιο και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια πολύ πιο επικαιροποιημένη αξιολόγηση της κατάστασης, καθότι γίνεται πιο ανησυχητική. Ε, μια νέα δεσμή μέτρων για τη μετανάστευση, από ό,τι φαίνεται, θα παρουσιάσει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε αυτή να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, πραγματικά στοιχεία. Αλλά ακόμα και η απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειε. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί και να δημοσιευθούν οι εκθέσει εφαρμογή. Δεν περίμεναν τόσο εντυπωσιακό αυτό που είπα <laughs> για να πέσει το φω. Gaslight ονομάζεται. Πάντως ε, τον Ιούλιο του 2017 λογικά θα έπρεπε να είχαμε λάβει τις ε, εκθέσεις ε, εφαρμογής όσον αφορά την οδηγία για το άσυλο, για τις συνθήκες υποδοχής. Θα έπρεπε επίσης να έχουμε μια έκθεση όσον αφορά το Δουβλίνο 3 και θα έπρεπε επίσης να έχουμε και μια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για το Eurodac. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τις νομικές αυτές υποχρεώσεις προκειμένου να έχουμε πραγματικά ένα σύμφωνο το οποίο να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η κυρία Ταρντίνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της μετανάστευσης. Ε, ελευθερία, δημοκρατία, ε, ανεξαρτησία, δημοκρατία, όχι ΙΣΙΑ, συγγνώμη. Έκανα λάθος. Ναι, ναι, συνεχίστε, συνεχίστε. Λάθος ε, την ομάδα σας έκανα. Έλεγα, Πρόεδρε, ότι μιλήσατε για μεγάλες επιτυχίες ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης αυτή την πενταετία. Τονίζοντας την ανάγκη να μην γυρίσουμε πίσω σε αυτό που ήταν παλιότερα η πολιτική για τα Στην πραγματικότητα, επίτροπε, η πραγματικότητα απέχει από αυτά που είπατε. Την πενταετία αυτή βιώσαμε όχι μόνο σοβαρά γεγονότα που επηρέασαν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιστών. Η ίδια η ασφάλεια αυτή αμφισβητείται κάθε μέρα από, την, από το συνεχιζόμενο φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης που δυστυχώς η Επιτροπή δεν, δεν μπόρεσε να περιορίσει. Μετά από πέντε χρόνια μπορούμε να πούμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό απέτυχε. Η παράτυπη μετανάστευση και το άσυλο απαιτούν εδώ και χρόνια μια απάντηση από την Ευρώπη που δεν καταφέραμε ωστόσο να δώσουμε διότι επιβάλαμε ε, υπερβολικά μεγάλο βάρος τα, στις ε, παραμεθόριες χώρες Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα που χρειάστηκε να ζητήσουν ελεημοσύνη βοήθεια από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. μα. ανησυχεί ιδιαίτερη κατάσταση στην Μεσόγειο, κατάσταση που είδε να μειώνεται ο αριθμό των νεκρών όντω όπω αναφέρθηκε, όχι ωστόσο λόγω του έργου που έκανε η Επιτροπή, αλλά του έργου που έκανε η μεταναστευτική πολιτική του Υπουργού κ. Σαλβίνη στην Ιταλία. Και τούτο επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Σε λίγε μέρε μετά την εγκατάσταση τη νέα ε, τριπλασιάστηκαν οι αφήξει. Ε, φοβόμαστε λοιπόν ότι πραγματικά η πολιτική που προωθείται αυτά τα χρόνια και ιδίως πρόσφατα ε, που και επανέρχεται πρόσφατα ε, μετατρέπει εκ νέου την Ιταλία σε στρατόπεδο προσφύγων της Ευρώπης. Εσείς είπατε ότι θα θέλετε να ξαναδείτε το Δουβλίνο. Η Επιτροπή έκανε μία πρόταση το 2016. Ρωτώ Επίτροπε, τι έκανε η Επιτροπή, τι θέλει να κάνει εάν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ζητηθεί. Ευχαριστώ. Το ECR. Ο κύριος Προκατσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρία ερωτήματα. Γρήγορα Πρώτον, πριν λίγες μέρες ο Γερμανός Υπουργός κ. Ζέχοφερ αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τη δημιουργία ενό προσωρινού μηχανισμού κατανομής των μεταναστών που εξετάζει και η συμφωνία αυτή θα επικυρωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Ένα είδος ευρωπαϊκού συστήματος που προβλέπει τις αφήξεις και, είναι λιγότερο, και καθιστά λιγότερο δεσμευτική και επίγουσα τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Με αυτή τη συμφωνία η Μάλτα και η Ιταλία θα έπρεπε να δώσουν τα λιμάνια του σαν ασφαλείς λιμένες αποβίβασης. Η Γαλλία και η Γερμανία θα παράσχουν με την πλευρά τους ε, ε, την, την εξέταση των ετοιμάτων και μέσα σε ένα μήνα θα μπορούσε να δοθεί απόφαση ή όχι για την προστασία. Πώς άλλαξε, γιατί άλλαξε έτσι ξαφνικά η στάση της Γαλλίας και της ε, Γερμανίας έναντι της Ιταλίας και της Μάλτας, κυρίως της Ιταλίας. Δεύτερη γρήγορη ερώτηση. Πριν λίγες μέρες είπατε Τι άτομα όπω η κυρία η Καρόλ Ρακέτε ε, προωθεί, την, ε, προωθεί ευρωπαϊκές και ηθικές ατομικές αξίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάζονται οι νόμοι. Τρίτον, η Όλαφ άρχισε μια έρευνα για το σύστημα υποδοχής των προσφύγων στην ε, Ιταλία γιατί από ό,τι φαίνεται πίσω από το σύστημα αυτό κρύβεται το οργανωμένο έγκλημα. Έχετε κάποιες πληροφορίες ε, σχετικά. Ευχαριστώ. Και η κυρία Έντ για την ΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Συνοτική Αριστερά για την εργασία που έχετε κάνει, μόλον ότι μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα. Νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί την ε, δική μα θέση από τη δικιά σα είναι ότι τα τελευταία πέντε χρόνια τα οποία ήταν και τα πιο δύσκολα χρόνια που έχουμε αντιμετωπίσει στον τομέα της μετανάστευσης από ιστορικής πλευράς, αν δούμε όλους αυτούς οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια, δεν μπορούμε απλώς να μιλάμε για συνέπειες και επιπτώσεις ε, όταν αξιολογούμε την κατάσταση. Νομίζω ότι κάποιοι θα πρέπει να πάνε στη φυλακή, ότι θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιε ποινικέ συνέπειε για το όσα συνέβησαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Εμεί πιστεύω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Αν δούμε την κατάσταση στη δική σα τη χώρα, την Ελλάδα, αν δούμε πώ έχει κατάσταση στα hot spot για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, σαφώς εκεί εξακολουθούν και υπάρχουν προβλήματα. Πάντως, δύο πράγματα θα ήθελα να γνωρίζω από εσά. Πρώτον, Πώς θα πρέπει να γίνονται δεκτοί οι μετανάστες, τι σύστημα ακολουθείτε, κάποιοι πάνε στη Γερμανία, κάποιοι σε άλλες χώρες, από τι εξαρτάται τελικά αυτό, σε ποια χώρα τελικά θα καταλήξουν. Από τη μία μέρα στην άλλη οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν τελικά τι τους επιφυλάσσει η μοίρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ποια θα είναι η δική σας συστάση και πώς θα κινηθεί επ' αυτού και το Συμβούλιο. Δεύτερον, αναφερθήκατε σε 320.000 Σύρους πολίτες οι οποίοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη χώρα τους μολονότι είχαν έγκυρα έγγραφα ταξιδίου. Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν μέσω της Τουρκίας, από την Τουρκία προς τα πίσω. Εμείς γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Δίνουμε τεράστια ποσά αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και δεν φαίνεται να ασχολούμεθα εν συνεχεία με την τύχη των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε ότι η χρηματοδότηση που δίνουμε στην Τουρκία τελικά δεν χρησιμοποιείται σωστά. Ποια είναι η δική σας η άποψη για τη στάση που έχει κρατήσει η Τουρκία απέναντι στους πολίτες αυτούς. Κύριε Επίτροπε, 20 ακόμα μέλη θέλουν να πάρουν το λόγο, επομένως θα πρέπει να είστε και εσείς σύντομος ε, στις απαντήσεις σας, προκειμένου να μπορέσω να τους δώσω έπειτα το λόγο. 10 λεπτά σας δίνω κύριε Επίτροπε, σας ζητώ να είστε λίγο ευσύνοπτος προκειμένου να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Είναι πολλά τα 10 λεπτά, θεωρείτε. 8 λεπτά, κύριε Επίτροπε, γίνεται να απαντήσετε μέσα σε 8 λεπτά. Ναι. Θα προσπαθήσω. Πάντως θα ήθελα να είναι επικοδομητική στάση μου στην όλη αυτή συζήτηση. Προφανώς δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ πέρα να δικαιολογήσουμε και να αιτιολογήσουμε την πολιτική μας. Ακολουθήσαμε μια πολύ ρεαλιστική στάση εξ αρχή, αντιμετωπίζοντα πολύ δύσκολε καταστάσει. Σα είπα εξ αρχή ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με τα κράτη-μέλη. Αφού όμω θέλετε να σα πω περισσότερα πράγματα, πρέπει να πω ότι κάποια προβλήματα αντιμετώπισα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντω, εν τέλει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα περήφανο γιατί είναι αυτό το οποίο υποστήριξε περισσότερο από όλους τη δική μας την πολιτική. Αυτή η πολύ στενή συμμαχία που υπήρξε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδήγησε τελικά στα πολύ θετικά αυτά επιτεύγματα και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σε μια εντελώ διαφορετική κατάσταση από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Και δεν αναφέρουμε μόνο σε αριθμητικά δεδομένα. Έχει αλλάξει πραγματικά η κατάσταση και η κοινοτροπία Και σε σχέση με αυτό που είπε η Ρομπέρτα, προφανώ θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Όσον αφορά το μέλλον, εναπόκειται στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει την πολιτική που θα ακολουθήσει. Πολύ σύντομα θα συναντήσετε τους νέους υποψήφιους επιτρόπους, θα συζητήσετε μαζί τους για τον δρόμο που θα ακολουθήσετε. Είναι κοινό αν θέλετε το έργο και κοινή ευθύνη για να καταφέρετε να σώσετε περισσότερες ζωές, να προστατεύσετε καλύτερα τα σύνορά μας και να δημιουργήσετε τελικά μια στρατηγική η οποία θα είναι πολύ πιο ανθεκτική, μια στρατηγική η οποία θα ταινίσει μάλιστα και το μέλλον και τι μελλοντικέ προκλήσει. Γιατί η μετανάστευση θα απασχολήσει και το επόμενο και το μεθεπόμενο κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να ασχοληθούμε και με το ζήτημα τη ασφάλεια, κρατώντα όμω τα δύο αυτά ζητήματα σαφώ ξεχωριστά. Μπορεί να υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ μετανάστευση και ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τι δύο αυτέ έννοιε, πράγμα το οποίο κάναν ορισμένε πολιτικέ ομάδες στην Ευρώπη, λέγοντας ότι η μετανάστευση αποτελεί όχημα για τρομοκρατία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι υπέτη τρομοκρατικών πράξεων στην Ευρώπη δεν ήταν μετανάστες. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Επομένως θα πρέπει να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα αυτά ξεχωριστά. Όσον αφορά το ερώτημα το οποίο θέσατε, Ρομπέρτε, για την κατάσταση στη Μεσόγειο, το είπα πολλές φορές στο παρελθόν ότι θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τις προσωρινές διευθετήσεις, το συντομότερο δυνατό. Και γι' αυτό το λόγο χαιρετίζω την πρόσφατη εργασία που ξεκίνησε μεταξύ των κρατών μελών ως προς αυτό. Είναι πολύ νωρί όμω για να καταλήξουμε σε κάποιες εκτιμήσεις, πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα όπως και στο παρελθόν, είναι έτοιμη να υποστηρίξει χρηματοδοτικά και επιχειρησιακά τις προσωρινές αυτές διευθετήσεις μέσω μάλιστα και των ευρωπαϊκών οργανισμών θα είμαι στη Μάλτα την επόμενη εβδομάδα εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Υπουργική Συνδιάσκεψη που θα λάβει χώρα με κάποια κρατημέλη, όχι με όλα. Πάντως το ζήτημα αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθεί και από όλα τα κρατη στο επόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων, όπου θα δοθεί μάλιστα και η ευκαιρία στους αρμόδιους υπουργούς να συζητήσουν το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να αποτελεί ένα μεταβατικό μέσο, αν θέλετε, αυτή η νέα προσωρινή διευθέτηση μέχρι να έχουμε και το νέο κανονισμό του Δουβλίνου. Πρόκειται λοιπόν για μια προσωρινή διευθέτηση η οποία θα βασίζεται σε θελούσια βάση και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει οποιαδήποτε νομοθεσία ή μελλοντική νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσει οποιαδήποτε διευκρίνηση πρέπει να δοθεί στο μέλλον για τον κονισμό του Δουβλίνου. Η απάντηση η λίστα πρέπει να είναι σφαιρική, ολιστική και θα πρέπει να προέλθει μέσω του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Και Ρομπέρτα, αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι εν είδη συμβουλής, ότι είναι πολύ καλύτερο να συνεργάζεστε μεταξύ σας, να συμμερίζεστε κοινέ αξίες ως προς την ακολουθητέα πολιτική και να μην ακούτε τις κυβερνήσεις σας και την πολιτική ηγεσία αναγκαστικά, γιατί περισσότεροι από αυτούς ουσιαστικά κοιτάνε προς τα πίσω, δεν ατανίζουν το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε εκπροσωπώντας Ευρωπαίους πολίτες να φέρουμε εις πέρα στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά πρέπει να πω και απευθύνομαι στον κύριο Κλοντ Μοράς ότι ήσασταν ένας πολύ καλός φίλος και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Όπως είπα στο λόγο μου, η νόμιμη μετανάστευση αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο μιας σφαιρικής πολιτικής για τη μετανάστευση. Η νόμιμη μετανάστευση δεν αποτελεί απλώ μία δική μου, θέλετε, πολιτική προσέγγιση. Είναι και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε επί τη ουσία. Θέλουμε την κινητικότητα, θέλουμε την κινητικότητα των πολιτών, αυτή πρέπει να προωθήσουμε και οι μελλοντικοί ιστορικοί θα χαρακτηρίσουν την εποχή μα ω την εποχή τη ανθρώπινη κινητικότητα. 500 εκατομμύρια άνθρωποι παντού στον κόσμο κινούνται αυτή τη στιγμή, αλλάζουν χώρα, ταξιδεύουν προκειμένου να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και μια εκτακτή συνδιάσκεψη για το ζήτημα αυτό. Σε ευρωπαϊκό παντός επίπεδο πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική στρατηγική για το μέλλον. Σοφίν Βέλτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια συλλογική μας αποτυχία να αντιμετωπίζουμε ακόμα ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν και χάνουν πολλές φορές τη ζωή τους. Όπως είπα και στο παρελθόν και θα το θυμάστε, δυστυχώς δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσει στο πλαίσιο της επεξεργασίας της σχετικής οδηγίας. Πάντως, παρόλα αυτά, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα όσον αφορά τις θεωρήσεις. Από τη δική μας την πλευρά συνεργαστήκαμε και με τις Ηνωμένε Πολιτείε και επιταχύναμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να βοηθήσουμε τα πέντε κράτη-μέλη να αποκριθούν στο πρόγραμμα απαλλαγής από τις θεωρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα ήμασταν σε επαφή και με τον ειδικό Διπραγματευτή των Πολιτείων και το βασικό ζήτημα, το πιο ακαθόδε ζήτημα ήταν η ασφάλεια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τώρα από την άλλη θα προσδώσουν σε αυτά τα πέντε κράτη-μέλη μία τεχνική, πρακτική καθοδήγηση για να αποκριθούν σε απαιτήσει αυτέ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν δεσμευθεί να υποδεχθούν στο πρόγραμμα αυτό απαλλαγή από τι θεωρήσει τα πέντε αυτά κράτη-μέλη, αυτή τη στιγμή τηρήσουν ή ανταποκριθούν μάλλον στι απαιτήσει που προκύπτουν από την Αμερικανική νομοθεσία. Και τα πέντε αυτά κράτη-μέλη έχουν σημειώσει απτή πρόοδο και πολλά από αυτά βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο να πληρούν πλήρω τα κριτήρια αυτά. Σύμφωνα με την αρχή τη αμοιβαιότητα, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη, και το τονίζω αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συνέπειες της αναστολής του καθεστώτος αυτού για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Επομένως, είμαστε κι εμείς έτοιμοι να εγκρίνουμε μια κατεξοδότηση πράξη αν έχουμε την κατάλληλη πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην οπισθοδρομήσουμε και να μην επιδεινώσουμε την κατάσταση από τη μία και την άλλη πλευρά. Τα αποτελέσματα που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον Καναδά αποδεικνύουν ότι μπορούμε να έχουμε μια πλήρη αμοιβαιότητα όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων μέσω τη κοινή προσήλωση, τη δέσμευση και των τακτικών διπλωματικών επαφών. Και είμαστε πεπισμένοι ότι οι προσπάθειέ μα θα ευδοκιμήσουν και ότι όντως θα καταφέρουμε να φέρουμε και τα πέντε αυτά κράτη-μέλη στο πρόγραμμα αυτό απαλλαγής από τις θεωρήσεις. Κυρία Τρίκ, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που μπορώ για πρώτη και τελευταία φορά να αντελάσω αυτές τις σκέψεις μου μαζί σας. Α μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας είναι μια συμφωνία μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και εμεί ε, ταχθήκαμε υπέρ τη πρωτοβουλία αυτή γιατί είχε θετικά αποτελέσματα. Η κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με, σε σχέση με κάποια χρόνια. Το 2016, μην ξεχνάμε ότι σε καθημερινή βάση είχαμε χιλιάδε πρόσφυγε οι οποίοι διερχόντουσαν, περνούσαν από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ο αριθμό αυτό έχει μειωθεί αυτή τη στιγμή και είναι πολύ πιο διαχειρίσιμος και Προσπαθούμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτικά να ενισχύσουμε τις ελληνικές αρχές αλλά και τις αρχές άλλων χωρών. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα. Η δήλωση αυτή, γιατί η δήλωση είναι, δεν είναι συμφωνία. Αν ήταν συμφωνία σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο, θα έπρεπε να είχε εγκριθεί, να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια και στην περίπτωση αυτή και θα έπρεπε επίση να έχει δώσει και τη σύμφωνη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα είχαμε καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο. Βρήκαμε λοιπόν, αν θέλετε, την πλατφόρμα αυτή, τη μέθοδο τη δήλωση που λειτουργεί στην πράξη. Τώρα, η δήλωση αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ω διαπραγματευτικό εργαλείο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει δώσει αποτελέσματα. 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και εμείς υποστηρίζουμε την Τουρκία προς αυτό. Τα χρήματα δεν πάνε στην Τουρκία. Τα χρήματα πάνε στο UNHCR, καθώς επίσης και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι οποίοι κάνουν εκεί πέρα μια εξαιρετική εργασία. Συνεπώς, θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο την συνεργασία αυτή. Τώρα, το αν είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία ή όχι αυτό σχετίζεται με τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων το τι γίνεται στην περιφέρεια, το οποίο ισχύει, το τι γίνεται στρατηγικά, γεωπολιτικά στην περιφέρεια δεν έχει να κάνει με την πολιτική της Ένωσης. Έχω και ένα κατάλογο εδώ, θα, απαντήσω πιο μετά. Μια σύντομη επιπλέον ερώτηση σε αυτή τη δήλωσή σας. Ο κ. Σαβραμόπουλο είπε, ξέρετε τι γίνεται, ότι το θέμα τη περιφέρεια της Τουρκία έχει γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Αλλά δέχεται ότι αν Σύριοι πρόσφυγε επιστρέφονται τώρα στη Συρία, αυτό σημαίνει επαναπροώθηση. Οι Σύριοι δεν, επαναπρο... δεν στέλνονται πίσω στη Συρία. Οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί που μπαίνουν στην Τουρκία και στην ε, Ευρώπη πρέπει να επιστραφούν. Κάποιοι θα έχουν διεθνή προστασία και κάποιοι όχι. Κοιτάξτε να δείτε, ο Επίτροπος παρουσιάζει τις απόψεις του. Ο μόνος τρόπος για να το χειριστούμε, έχουμε 20 συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν, ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε πειθαρχημένοι. Ένα λεπτό καθένας. Δεν γίνεται αλλιώ. Και έχουμε και ένα περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Ένα λεπτό παρακαλώ. Μη με υποχρεώνετε να ασκώ τις εξουσίες του Προέδρου χτυπώντας ένα λεπτό, μία ερώτηση. Τέλος. Ξεκινούμε τον κύριο Πίτενς, ο οποίος ζήτησε να είναι πρώτος γιατί θέλει να φύγει. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την εξαιρετική δουλειά του. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση έχω για την ε, κοινή δήλωση με την Τουρκία. Η επιστροφή από την Τουρκία στην, από Ελλάδα Τουρκία δεν λειτουργεί. 95 άτομα α, φέτος μόνο. Ο χαμηλότερος αριθμός επιστροφών σε σχέση με το ξεκίνη, από το ξεκίνημα της ε, κοινή δήλωση. Πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των επιστροφών στην Τουρκία από την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, σύμφωνα με το Human Rights Watch, μια γυναίκα έχει, γυναίκες αναφέρουν συχνές ε, σεξουαλικές παρενοχλήσεις στα hot spot στην Ελλάδα. Τι διαδικασίες ακολουθεί η Επιτροπή για την εξασφάλιση των γυναικών και των ασυνοδεύτων ανηλίκων. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των ομάδων υποστήριξης της Ένωσης για τα θέματα ασφάλειας γυναικών και ανηλίκων στα hot spots και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού γενικά. Στάνη. Ασμάνη. Διορθώνει το όνομα. Ευχαριστώ τον κύριο Ευραμόπουλο. Στην κοινή δήλωση θα αναφερθώ κι εγώ. Το θέμα είναι να αποφύγουμε την παράτυπη μετανάστευση και να διευκολύνουμε και να μειώσουμε την ανθρώπινη τραγωδία. Αυτό μπορεί να είναι ένα παράδειγμα για το μέλλον. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι έχει κάνει εν μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδίω για την Τουρκία πιστεύω ότι δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα από μία χώρα ένα μηχανισμό. Δεν είναι χρήσιμο αυτό. Επίσης, τι άποψη έχετε για τις ε, πρόσφατες δηλώσεις και απειλές του Ερντογάν ότι θα στείλει πρόσφυγες ε, στην Ένωση και ότι η Τουρκία δεν δέχεται πλέον πρόσφυγες, επιστροφή προσφύγων από την Ελλάδα. Τι δράση λάβατε για τον τομέα αυτό. Φόιδο. Καλησπέρα. Δεν θα υποβάλω ερώτηση, θα εκφράσω την αναγνώρισή μου προς τον Επίτροπο. Εκ πρώτης, ε, από πρώτο χέρι μπόρεσα να βιώσω την μεταναστευτική κρίση. Τέτοια μεταναστευτική πίεση είχε δεκαετίες να βιώσει η Ευρώπη. Παρά, παρότι ωστόσο Πολλά κράτη-μέλη δεν το πίστευαν. Εσείς αντιμετωπίσατε ουσιαστικά το ζήτημα και προσπαθήσατε να βρείτε λύση που θα ανταμοκρίνονται στην πραγματικότητα της Μεσηγείου. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να εκφράσω την αγνώρισή μου για την προσπάθεια και τη δουλειά σας. Τη δουλειά σας για τη βελτίωση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την μετανάστευση και το άσυλο ήταν επιθυμία σας να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ όλων των κρατομελών για να υπάρξει ένα κοινό σύστημα ασύλου. Δεν κατέστη δυνατό, αλλά δεν κατέστη δυνατό όχι διότι δεν προσπαθήσατε εσείς. Τελειώνω πρόεδρε, πρόεδρε ευχαριστώντας τον κύριο Αβραμόπουλο για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εύχομαι ό,τι καλύτερο στι νέες, στις νέες του στον κύριο Επίτροπο. Πόλας, πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για αυξημένο επίπεδο ασφάλειας στα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό που με ανησυχεί είναι η υλοποίηση αυτής της ασφάλειας, διότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες και για την νόμιμη μετανάστευση, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ασφάλειας. μεταξύ Βοσνίας και Κροατίας περνάει συνεχώς κόσμος παράτυπα. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν καταστάσεις όπου ε, διαπιστώσαμε μεταξύ των δύο αυτών χωρών από την Κροατία συλλογικές ε, απελάσεις. Τι ε, τακτικά μάλιστα, όχι μόνο μία φορά, τι μέτρα λαμβάνονται για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η πρώτη μου ερώτηση διαρωτώ με αν μπορείτε να μας πείτε τι αποδείξεις έχετε για να βασιστείτε ε, στο θέμα ότι ε, υπάρχει αυτή η τρομοκρατία ή δεν υπάρχει, συνδέεται η μετανάστευση αυτή με πράξεις τρομοκρατίες. Μερικές εταιρειε δεν, εταιρείες δεν συνεργάζονται εθελοντικά. Οι διάφορες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το νομοθετικό καθεστώς. Η ε, κυρία Ιντεβάλντ είπε ότι η Europol ε, θέλει ε, για ε, το θέμα αυτό της, των δεδομένων. Έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Κύριος Παπαδάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Αβραμόπουλε, δηλώσατε περήφανος και μίλησατε για κληρονομιά. Την Παρασκευή πήγα στη Μόρια. 10.500 πρόσφυγες, ένας γιατρός, ένας παιδίατρος. 4.000 σε σκηνές. 3.000 στη Σάμο επίσης σκηνές. Το ερώτημα ένα. Ο χειμώνα θα βρει τους πρόσφυγες σε αυτή την κατάσταση. Έχετε σχεδιασμό πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα τώρα. Και δεύτερο ζήτημα. Το επιχείρημα ήταν ότι η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σταματάει τις ροές. Αυτό έχει καταρριφθεί. Ποιος ο λόγος λοιπόν συνέχισης και του απαράδεκτου καθεστώτος των hot spot και της δήλωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Господин Комисар, благодаря за съвместната ни работа Ο κύριος Ράντεφ, αντιπρόεδρος κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, μέσα σε μια μέρα στη Λέσβο, πάνω από 600 άτομα φτάσαν από την Τουρκία. Και παράλληλα, ο Ερντογόν τι τελευταίε μέρε έχει πει ότι θα ανοίξει τι πύλε τη Τουρκία και ότι θα κατακλείσει κατά αυτόν τον τρόπο με πρόσφυγε και μετανάστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν δώσει περισσότερα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μα είπε. Τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη Λέσβο πρέπει να μας απασχολήσουν, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια νέα κρίση σαν αυτή του 2015. Ο κύριος Ρομπέρτη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την πολύ θετική συνεργασία που είχαμε και το εκτιμήσαμε αυτό επίσης και στη συνάντηση που είχαμε μαζί σας στην Ιταλία όταν ήμουν γενικό αγγελέα κατά τη μαφία στη χώρα μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την έντονη δέσμευση και προσήλωσή σα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είχαμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία και εσείς ευχόσασταν, αλλά τουλάχιστον ξεκινάμε όπως είπατε από μια θετική βάση. Ως προς αυτό λοιπόν σας θέτω δύο ερωτήματα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι θέλουμε να φτάσουμε σε μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών που συμμετέχουν εθελουσίως. Εσείς είπατε ότι πρέπει να έχουμε ένα βιώσιμο μηχανισμό αλληλεγγύης. Όμως ποια προβλήματα πιστεύετε ότι θα έχουμε, ποιες δυσκολίες ενδεχομένως να προκύψουν, οι οποίες θα μπλοκάρουν αυτό το μηχανισμό, τον εθελούσιο της αλληλεγγύης. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό σε σχέση και με το σκάφος Ocean Viking, το οποίο έχει πλησιάσει τις ακτές της Ιταλίας. Δεύτερον, τι θα γίνει με τους πρόσφυγες εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, στα hot spot. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ε, επιχειρήσεις όπως η Σοφία, η Γιουναφόρ ή άλλες επιχειρήσεις στο παρελθόν αποτελούν πάρα πολύ συχνά μόνο αποστολές παρακολούθησης. Δεν πιστεύετε ότι οι άλλες επιχειρήσεις στο παρελθόν αποτελούν πάρα πολύ συχνά μόνο αποστολές παρακολούθησης. Δεν πιστεύετε ότι η επιχείρηση Σοφία θα πρέπει να ξεκινήσει με συγκεκριμένα σκάφη και να μπορεί πραγματικά να επεμβαίνει αποτελεσματικά στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δύο ερωτήσεις. Ε, στην αναθεώρηση του πακέτου ασύλου, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο προχώρησαν μαζί. Αυτό που μπλοκάρει είναι το Συμβούλιο. Η ιδέα που διατυπώθηκε από μερικούς να ξαναρχίσουμε όλη την εργασία με μια νέα πρόταση της Επιτροπής μας φαίνεται στήρα το να ξαναρχίσουμε από μηδενική βάση. Τι δρόμο βλέπετε, τι μέσο για να ξεμπλοκάρουμε την εργασία ή την οικοδόμηση μιας λύσης μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ουγγρικά. nemzeti hatáskör. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη αναγκαστικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μην ξεχνάμε ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα ζήτημα, ζήτημα εθνικής αρμοδιότητος. Νομίζω ότι αντί να ασκείτε πίεση θα ήταν καλύτερο να προβληματιστείτε λίγο για τα βαθύτερα αίτια και ουσιαστικά να προστατεύουμε καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε για ποιο λόγο ξεκινούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύουμε καλύτερα τα εξωτερικά μα σύνορα, όπω και η Ουγγαρία προστάτευσε αποτελεσματικά τα νότια σύνορά τη. Νομίζω ότι ο έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο προστασία τη Ευρώπη και θα πρέπει να τροποποιήσουμε την, πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση και να προστεύουμε καλύτερα τα εξωτερικά μα σύνορα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε εκατομμύρια ανθρώπους από τον έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, θα τους δώσουμε ένα κίνητρο για να έρθουν εδώ και νομίζω ότι αυτό αντιτίθεται στην πραγματική θέληση των Ευρωπαίων και στις πραγματικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Μία ερώτηση για το, για το Δουβλίνο δεν μπορώ να μην την κάνω. Δική σας, δικό σας δημιούργημα νομίζω ήταν. Πώς θα προχωρήσει, πιστεύετε, η συζήτηση για αυτή την κρίσιμη μεταρρύθμιση. Θα, θα καταφέρει το Συμβούλιο να βρει λύση. Η αλλαγή, πιστεύετε ότι η αλλαγή της κυβέρνησης στην Ιταλία θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος ή πιστεύετε ότι η Επίτροπη σκέφτεται να αποσύρει την πρόταση και να υποβάλει νέα. Τώρα, το όλο αφήγημα για τη μετανάστευση, το οποίο είναι ένα στρεβλό αφήγημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Η εικόνα που προέρχεται είναι μια υπερβολικά αρνητική εικόνα. Έχει γίνει προσπάθεια από πλευράς κομισιών να δώσει μια θετική παράμετρο της μετανάστευσης. Δεν πρέπει και η Επιτροπή να κάνει μια πολιτική επικοινωνιακή που θα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Μάρκαντ. Γερμανικά θα μιλήσω. Ευχαριστώ. Μας είπατε ότι η λύση δεν είναι ε, να ε, στέλνουμε τα άτομα από την Τουρκία στην Συρία. Ο Ελντοάν είπε ότι είναι έτοιμος ε, να ξαναστείλει πίσω στη Συρία ένα εκατομμύρια Σύρους. δεν ξέρω, ψεύδεται. Ε, στην, ανάμεσα στα σύνορα Κροατίας και Βοσνίας γίνεται λόγος για το pushback, έτσι το ονομάζουν, ε, για το, για, και για αντιδράσεις βίας. Η Επιτροπή έχει γνώση της κατάστασης αυτής, της πυρήταδαποθήκης αυτής και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αυτό το σύνορο. Η Επιτροπή έχει γνώση των όσων γίνονται στην Μεσογειακή Λεκάνη όπου υπάρχουν οργανώσεις που προσπαθούν να βοηθούν άτομα αλλά που επίσης διονίζουν και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι η βασική μας αξία δεν είναι να προστατεύουμε την τάξη, αλλά να προστατεύουμε την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου όντως. Αυτή είναι η πολιτική μας η ουσία. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο θέμα που ήδη τέθηκε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η χρήση αυτού του pushback, του παράνομου από την Κροατία, από την συνοριακή αστυνομία, είναι κάτι το γνωστό εδώ και καιρό. Εδώ και ε, μερικές εβδομάδες η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά. Σύμφωνα με τις ε, ΜΚΟ ε, δεν έχουν φτάσει στην Μπίχατς τα κονδύλια. Κάπου σταμάτησαν αυτά τα κονδύλια, κάπου μπλοκαρίστηκαν. Είναι 800 πρόσφυγες που προβλέπεται ε, να μείνουν εκεί. Η κατάσταση είναι δραματική. Στην Βοσνία Ερζεγοβίνα η κατάσταση στην Μπουτσάκ ε, θέτει ε, κινδύνους ασφάλειας για αυτούς που έχουν επανεγκατασταθεί. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να διορθώσει αυτήν την κατάσταση, πώς μπορεί να υποστηρίξει τις ΜΚΟ και τους εθελοντές που εργάζονται στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος η κυρία Φεράρα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο για την δουλειά, για το έργο που έχει κάνει σε μια δύσκολη και ευαίσθητη θέση με πολλές ε, δυσχέρειες, το είδαμε Είχαμε, παντ, είχαμε μερικές φορές συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια πολύ καλή και έντιμη συνεργασία για να πετύχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Και επανέρχομαι στο σημείο αυτό για τα ερωτήματά μου. Καταρχήν, καταρχάς, αφήξεις. Μπορεί να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία που διαφαίνεται μεταξύ κάποιων πρόθυμων κρατών μερών και που θα επικυρωθεί στη Μάρτα σε λίγες μέρες. Ε, στην πράξη θα είναι μια ενισχυμένη συνεργασία που δεν προβλέπεται αλλά και που βασίζεται στο άρθρο 80 της συνθήκης. Δεύτερον, με βάση την εμπειρία του μπορεί να είναι αυτό ένα... Τι, τι μπορεί να χρησιμοποιήσει για να πιέσει τα κράτη που δεν ενδιαφέρονται για την συμμετοχή αυτή, διότι στην πράξη υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης κάποιων κρατών μελών στη συνεργασία σε ό,τι αφορά την κατανομή των ευθυνών. Τρίτη ερώτηση, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς ήμασταν αντίθετοι με τη συμφωνία αυτή, ιδίως στον τρόπο λειτουργία της από agreement έγινε deal και μετά έγινε statement. Πέρασε, ε, εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο χωρίς να, να κριθεί και έγινε ένα νομικό εργαλείο που δεν έχει καμία νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συμφωνώ με τα όσα είπατε και πραγματικά επιδοκιμάζω τα όσα έχετε καταφέρει όσον αφορά τον χώρο του Σέγγεν. Το πρόβλημα που έχουμε όμως στο εσωτερικό του Σέγγεν αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε ελέγχου στα εσωτερικά μας σύνορα, μεταξύ των κρατών μελών δηλαδή. Το δικό μου το ερώτημα είναι το ακόλουθο. τι θα μπορούσε πραγματικά να μας βοηθήσει να σπάσουμε, να βγούμε από το διέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε και να επιστρέψουμε τελικά στην κατάσταση που βρισκόμασταν στο παρελθόν. Να έχουμε ένα βιώσιμο χώρο Σέγγεν που να λειτουργεί σωστά, χωρίς όμως εσωτερικού ελέγχους από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο χώρο Σέγγεν. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Βάσλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Είπατε ότι ε, είναι αναγκαίο να έχουμε μια εταιρική σχέση και συνεργασία με τρίτες χώρες. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το θέμα αυτό, ιδίω με την εταιρική σχέση που θα μπορούσαμε να είχαμε με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όσον αφορά τις ε, μεταναστευτικές ροές. Και ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ε, στην κατάσταση που έχει προκύψει στα σύνορα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ότι τα σχολιά τους δεν ήταν πάρα πολύ σαφή και πάρα πολύ ακριβή. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η δική σας η αποτίμηση όσον αφορά την συνεργασία αυτή και όσον αφορά την εφαρμογή της εταιρική αυτής σχέσης και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να είχαμε από μία υποστήριξη προς τη Βοσνία Ζεγοβίνη ή άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσον αφορά την αντιμετώπιση πάντα των μεταναστευτικών ροών και πώς μπορούν να ευοδοθούν οι προσπάθειες αυτές και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σλάντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δράτω με τις ευκαιρίες για να σα ευχαριστήσω προσωπικά για την πολύ θετική συνεργασία που είχαμε και για τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις συζητήσεις που είχαμε τότε. Μόλον δεν καταφέραμε να βρούμε τελικά μια σφαιρική λύση για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε πολλά ζητήματα και καταφέραμε να αλλάξουμε τα πράγματα όσον αφορά τον κανονισμό Δουβλίνο 4. Βλέπετε όμως ότι μπορεί να άλλαξα θέση και αρμοδιότητες, πάντως το ζήτημα αυτό της μετανάστευσης και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων θα εξακολουθεί να αποτελεί ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές για μένα. Συμφωνώ τα όσα είπατε για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και είναι σαφές ότι είναι ανθρώπινο καθήκον μας να διασώσουμε ζωές στην Μεσόγειο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για να απαγορεύσουμε στους ανθρώπους να επιβιβάζονται σε σκάφη τα οποία μπορεί να τους οδηγήσουν τελικά και στον ίδιο το θάνατο. Νομίζω ότι όσο υπάρχουν κίνητρα, όσο διαφαίνεται η ευκαιρία να καταφέρουν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξακολουθήσουν να επιβιβάζονται στα σκάφη αυτά. Αν μπορούσατε να επιστρέψετε στο παρελθόν, θα αλλάζατε εντελώ τη στάση για κάποια ζητήματα, τι θα κάνετε διαφορετικά. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα προκειμένου να δώσουμε αντικίνητρα στου ανθρώπου να επιβιβάζονται στα σκάφη αυτά. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τι ε, χώρε τη Αφρική και να ενημερώσουμε καταλήλω του ανθρώπου αυτού για το πώς νομίμως μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ούριτσε παρακαλώ. Ο κύριος Ούριτσε είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ που τη θέση αυτή, γιατί νομίζω ότι είστε υπεύθυνο ουσιαστικά και για την παρακμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κλείνουν οι εκκλησίες, αυξάνεται η τρομοκρατία παντού στην Ευρώπη και πολλά άλλα δεινά αντί να αποτρέπει την παράνομη παράτυπη μετανάστευση, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα πάντα για να προωθήσει αυτή τη μετανάστευση. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να το δει αυτό και βλέπω ότι θέλετε να δημιουργήσετε μόνιμα συστήματα υποδοχής και ανακατανομής των μεταναστών. Ελπίζω πραγματικά να ξυπνήσουμε σύντομα στην Ευρώπη και να μην υποστηρίζουμε πλέον πολιτικούς οι οποίοι προδίδουν την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέ έχει το λόγο. Κύριε Αβραμόπουλε, τον Δεκέμβριο 2017 είχατε ένα άρθρο με τίτλο «Οι μετανάστες είναι εδώ για να μείνουν, πρέπει να ρυθμίσουμε τις πολιτικές μας ανάλογα. Αφήσατε ανοιχτές τις πύλες της Ευρώπης και επιτρέψατε ε, τις ροές. Ορμπάν ε, προτίμησε να προστατεύσει τα σύνορα. Εσείς αφήσατε ε, τους μετανάστες στη Μεσόγειο, στη Λιβύη. Ο Σαλβίνη τους σταμάτησε. Θέλετε να ανοίξετε την αγορά εργασίας στους πρόσφυγες ενώ πρέπει να δώσουμε θέσεις εργασίας στους πολίτες μας ενώ έχουμε ανεργία από τα κράτη-μέλη. Έχετε μια σύμπραξη με την Τουρκία του Ερντογάν δίνοντας 6 δισεκατομμύρια και εξακολουθεί σήμερα να εκβιάζει και ζήτησε ακόμη περισσότερα χρήματα ε, και ε, πύλησε να ανοίξει τις ε, πύλες προς την Ευρώπη. Βοηθήσατε λοιπόν την παράνομη, παράτυπη μετανάστευση και ο διάδοχός σας θα προστατεύσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής διότι αυτό η μετανάστευση επίσης ε, απειλεί την δική μας ταυτότητα. Ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Το λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος, κύριε Βδαμόπουλε. Well, let me start from a very political... Ας ξεκινήσω από μια πολύ πολιτική παρατήρηση. Αν η άκρα δεξιά με επενούσε γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν θα ήμουν ένα ευτυχή, ένας ευτυχής άνθρωπος. Αλλά είμαι ευτυχής Ευρωπαίος πολιτικός, διότι όλα αυτά τα χρόνια δούλεψα σκληρά μαζί σας, με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε εν τέλει να πούμε ότι κάναμε ένα βήμα μπρο. Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Θυμηθείτε όμως από πού ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια. Κάποιοι λείπατε, αλλά κάποιοι θυμάστε ότι η δουλειά δεν ήταν εύκολα. Εύκολη. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου, κάποιοι στην Επιτροπή με είχαν χαρακτηρίσει ατυχή, ε, άτυχο άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι μετά πέντε χρόνια μπορώ να πω ότι ήμουν ο τυχερότερος, διότι μπορούσα να πω ότι έκανα αυτό που είχα πει στην ακρόασή μου. Ευρωπαίος Επίτροπος που προστατεύει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεματοφύλακα των συνθηκών και των αξιών πάνω στις οποίες χτίστηκε η Ευρώπη. Και η Ευρώπη θα συνεχίσει να υπάρχει μόνο αν οι αρχές αυτές της αλληλεγγύης και της ευθύνης γίνονται σεβαστές από όλους μας, όλα τα θεσμικά όργανα, όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ήμουν λοιπόν ένας φανατικός Ευρωπαίος και είμαι περήφανος γι' αυτό. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Δεν θέλω να πω ό,τι είχα πει στην αρχή. Κύριε Κέλλερ, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε, ούτε πρέπει να ξαναγυρίσουμε ε, στο, στο μηδέν και να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Πολλά έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια. Ίσως χάρη στην μεταναστευτική κρίση και την κρίση ασφάλειας θα έπρεπε να είχαμε συνεργαστεί. Ο κύριος Ασμάνη και ο κύριος Πίτερς με ρώτησαν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα για τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται υπέρ της υλοποίηση της ε, δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που αποδίδει. Αυτό είναι μια δέσμευση αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαία ε, εφαρμογής απαιτεί προσπάθειε και από τι δύο πλευρέ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε γιατί απάντησα νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα ελληνικά νησιά, συνεργαζόμαστε στενά με τι ελληνικέ αρχέ. Η κατάσταση στην ΣΥΜ, στη ΣΑΜΟ και στη Λέσβο είναι ακόμα πολύ δύσκολη. Η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πλήρως να βελτιώσει, να, να προετοιμάσει καλύτερα τα νησιά για τον επερχόμενο χειμώνα και είμαστε μαζί τους, τους υποστηρίζουμε πολιτικά, οικονομικά και πρακτικά. Μια άλλη παρατήρηση, οι γυναίκες και τα παιδιά, οι ευάλωτοι μετανάστες, χρειάζονται την προστασία μας. Οι αρχές είναι υποχρεωμένες να αναλάβουν τα αναγκαία μέτρα. Σας υπενθυμίζω ότι είναι εθνική ευθύνη. Ο ρόλος της Ένωσης και της Επιτροπής είναι συντονιστικός και να παράσχει στα κράτη-μέλη, ιδίω της ε, πρώτης γραμμή υποστήριξη. Αυτό κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Υποστηρίζοντας τις χώρε που αντιμετωπίζουν πιέσει. Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεδομένα και, και, και καταγραφή δεδομένων. Ξέρω πόσο ευαίσθητη είσαι αυτό. Πριν εξετάσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή μια σχετική ε, νέα μελλοντική πολιτική, πρέπει να έχουμε πλήρη γνώση της κατάστασης και να περιμένουμε τις αποφάσεις των, των, τις αποφάσεις των δικαστηρίων που θα δώσουν ευκαιρία να διευκρινίσουμε περαιτέρω κάποια στοιχεία της τωρινής νομολογίας. Και το προγενέστερο και το Συμβούλιο υπογράφησαν τη σημασία να βρεθούν λύσεις. Εν τέλει, η νέα Επιτροπή θα έχει την ευθύνη να, εξετάσει τις εναλλακτικέ που υπάρχουν. Για τον κύριο Μπαρτόλο. Δεν μπορώ να προβώ σε εικασίες για τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής. Σύντομα θα ακούσετε τους επιτρόπους ε, και μπορείτε να τους ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Τώρα, για να πώς ξεμπλοκάρουν οι συζητήσεις για τα θέματα του ασύλου. Το είπα εισαγωγικά. Απαιτείται εμπιστοσύνη, που είναι βασικό σε όλους τους τομείς, όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και το μέλλον του Δουβλίνου. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, αμοιβή εμπιστοσύνη. Και ελπίζω στο μέλλον τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εμπιστεύονται το ένα το άλλο περισσότερο. Κύριε Χιλμπέκη, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να παίξουν πλήρω το ρόλο τους σε όλες τι πολιτικές μας. Αν έχουμε πολιτική θέληση, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με την υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος ασύλου, που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο μέλλον, διότι δεν ξέρουμε ε, τι μας περιμένει στο μέλλον. Όχι μόνο ε, για τα κράτη-μέλη της ε, Νότιας Ευρώπης. Η Ευρώπη περιτριγίζεται από έναν κύκλο αστάθειας από την Ουκρανία μέχρι την Τινησία τα ευρωπαϊκά σύνορα πρέπει να τύχουν καλύτερης προστασία. Αυτό έχουμε προσπαθήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη με τις πολιτικές και τους μηχανισμούς τους κατάλληλους. Αγαπητή Λάουρα, ε, αναφέρθηκα και προηγουμένως στο, στην συνάντηση που θα έχουμε τη Δευτέρα στη Μάλτα που ελπίζω να έχει θετικά αποτελέσματα. Κύριε Μπίλτσικ, ας μην ξεχνούμε ότι όλα τα, οι προσπάθειες, οι προτάσεις που θέσαμε επιτάπητος και που εφαρμόστηκαν ε, αποβλέπουν σε καλύτερη διαχείριση των κοινών εξωτερικών μας συνόρων. Άκουσα προσεκτικά τις παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων σας. Υπάρχει ένας κοινό παρανόμαστής, αλλά όλες τα πολιτικά κόμματα εδώ, οι ομάδες και τα κράτη ζητούν καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων, διάσωση ζώων, καλύτερη καταπολέμηση των διακινητών ε, και το τράφικινγκ ε, και την ε, και να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για το μέλλον, υιοθετώντα μια στρατηγική ολιστική για την μετανάστευση ε, και ε, την ασφάλεια. Έχουμε εδώ τα διάφορα δομοστοιχεία, τους πυλώνες που πρέπει να συμπληρωθούν στο μέλλον και θα είναι από τις βασικές προσπάθειες ε, της Μελλοντικής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου όσον αφορά το Σέγγεν. Ήμουν σαφή στην αρχή. Είναι καιρός να σταματήσουμε να ε, εξαλείψουμε τους εσωτερικούς ελέγχους και να υπάρξει καλύτερη ε, συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες μας. Ε, βεβαίως η νέα συνοριοφυλακή μπορεί να παίξει έναν πολύ ισχυρό ρόλο. Τώρα θα ήθελα να στραφώ προς τον Έλληνα φίλο μου, που έθεσε την ερώτηση ελληνικά και έτσι θα μπορέσω κι εγώ να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Δεν αμφισβητώ αυτό που είπατε, ότι πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες στα νησιά. Οι ελληνικές αρχές, το είπα και πριν, έχουν την πλήρη υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οικονομικά, επιχειρησιακά, πρακτικά. Αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί περίπου 750 στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθ' όλων το μήκος των, Ευρωπαϊ... των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Η οικονομική στήριξη της Ελλάδος έχει φτάσει στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά όπως είπα πρωτήτερα, η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες της, είμαι σε ανοιχτή γραμμή με την καινούργια ελληνική κυβέρνηση και θέλω να πιστεύω ότι όλα τα σημεία που θίξατε στο σύντομο χρονικό διάστημα που μένει μέχρι να ξεκινήσει ο χειμώνα και εμά μα ανησυχεί πάρα πολύ ο χειμώνα για να μην ξαναδούμε σκηνέ σαν και αυτέ που είδαμε πριν από δύο περίπου χρόνια στα νησιά. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Εμεί θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Σε ό,τι αφορά την ε, παρατήρησή σα και πάλι για την ε, ε, ευρωτουρκική συνεννόηση. Είναι δήλωση. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι συμφωνία. Τηρείται αυτή τη στιγμή. Αναγνωρίζουμε αυτό που είπαμε, ότι 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται εκεί και την χάνουν της στήριξης που απαιτούν και οι ίδιοι αλλά και υποχρεωμένοι η Τουρκία να δώσει με την δικιά μας οικονομική στήριξη. Θέλω να κάνω όμως μια διευκρίνηση. Επειδή αυτή η παρανόηση υπάρχει, τα χρήματα αυτά δεν δίνονται στην Τουρκία. Τα χρήματα αυτά δίνονται στους διεθνείς οργανισμούς και μάλιστα στα Ηνωμένα Έθνη, στον UNHCR και στον IOM που έχουν αναλάβει να καλύπτουν τις ανάγκες σε ιατρική περίπτωση σε φαγητό, σε καθαρό νερό και σε στέγαση όλων των ανθρώπων. Που όμως, επειδή είναι χαρακτηρισμένοι ως πρόσφυγες και θέλουν να μένουν εκεί γιατί ακριβώς είναι κοντά στα σπίτια τους έτσι ώστε όταν σε κάποια στιγμή λήξει ο πόλεμος στη Συρία να επιστρέψουν ε, στα χωριά τους και στις πόλεις τους. Είναι μεγάλος αριθμός. Υπολογίζεται σε 3,5 εκατομμύρια. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και 4 εκατομμύρια. Εκείνο που ελέγχθη όμως πρόσφατα και εμεί δεν είμαστε εδώ να ερμηνεύσουμε τις δηλώσει ε, του πρόεδρου της ε, Τουρκίας. Μπορούμε όμως να κατανοήσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ε, Τουρκία. Γι' αυτό και έχουμε ανοιχτό διάβλο συνεννόησης με την τουρκική κυβέρνηση πέρα και πάνω από τα άλλα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και επιλέξαμε αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο της δήλωσης για να συνεργαστούμε και να συνεννοηθούμε και να αναγνωρίζουμε τι συμβαίνει και αν αυτή η συμφωνία, αυτή η συνεννόηση αποδίδει. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον UNHCR και τον IOM για να προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε αυτούς τους ανθρώπους. Την άλλη μεριά όμως, θα ήθελα να σημειώσω κάτι άλλο. Από την ώρα που επιταχυνθούν στα ελληνικά νησιά, στα hot spots, οι διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων ασύλου θα είναι και πολύ πιο εύκολο να επιστρέφονται εκείνοι που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίες. Εμείς είμαστε δεσμε, δεσμευμένοι ως Ευρώπη από τη Σύμβαση της Γενέβης. Είμαστε εναντίον των pushbacks, το λέω για μία ακόμα φορά για να το ξεκαθαρίσουμε, και θα ήθελα να κάνω και μία ακόμα πολιτική παρατηρήση απαντώντας και σε κάποιους συναδέλφους των τελευταίων αρθρών έναν ακραίο πολιτικό λόγο. Δεν θα επιτρέψει αυτή η Επιτροπή μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας εδώ η Ευρώπη να γίνει φρούριο. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Και επειδή ξεχνάνε πάρα πολύ, θα ήθελα να του θυμίσω ότι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η φράση Fortress Europe ήταν από τον Χίτλερ το 1932. Η Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε αρχές και αξίες, δημοκρατικές αξίες και σε τελευταία ανάλυση καλό θα είναι να ξέρουν κάποιοι ότι οι ιστορικές ηγεσίες τους πήραν μια μέρα την απόφαση να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Γι' αυτό είπα πρωτήτερα αναφέρομαι σε κυβερνήσεις και όχι σε κράτη. Μόνο που φαίνεται ότι ξεχνούν οι κυβερνήσεις ότι έρχονται και απέρχονται. Και όταν κάποιες ιστορικές ηγεσίε μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού πήραν την απόφαση να εντάξουν τις χώρες στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεσμεύτηκαν να τιμούν, να υπηρετούν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές πάνω στις αξίες πάνω στις οποίες έχει στηθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που κάνω αυτόν τον καιρό ήταν να διαχειριστούμε την υπόθεση με πρακτικέ πολιτικέ που έδωσαν τα αποτελέσματα αυτά που όλοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν, γι' αυτό δεν είμαστε εκεί που είμαστε πριν, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που θέσαμε ως προτεραιότητα ήταν να είμαστε οι φύλακε των συνθήκων. Διότι χωρί τι αρχέ αυτέ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει. Και οι απαντήσει που σα έδωσα μέχρι τώρα σε αυτό κατατείνουν και αυτό εξηγούν πώ αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μα. Και γι' αυτό σα είπα ότι η Επιτροπή Juncker και όλοι εμεί που πλαισιώσαμε την προσπάθεια του ιδίου αλλά και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που μας ενεπιστεύτηκε αυτή την αποστολή ήταν να φέρουμε αποτελέσματα. Και κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν φέραμε αποτελέσματα. Τώρα, για εκείνους που δεν πιστεύουν σε αυτό, αυτό είναι απόλυτο δικό τους ε, δικαίωμα. Εξάλλου, είμαστε στον ναό της δημοκρατίας, αποκούνται διάφορες απόψεις. Αλλά μια παρατήρηση επιπλέον. Οι βασικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας, και μετανάστευσης, γιατί είναι και τα δύο αυτά θέματα μέρος του χαρτοφυλακίου που μου ανεπιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή, εκεί είχα τη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων που έχουν ταχθεί να υπηρετούν την ιδέα της Ευρώπης. Και είναι η συντριπτική πλειοψηφία που πιάνει σε αυτό το χώρο το 80 με 85%. Όταν έχεις πίσω σου λοιπόν όλε αυτέ τι δυνάμει προχωράς μπροστά. Αξιολογείσαι, κρίνεσαι, ενισχύεσαι, ενθαρρύνεσαι. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Επιτροπή αυτή, τη ΛΥΜΠΕ Κομίτη, για την οποία οφείλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Όταν επρόκειτο να εμφανιστώ για το hearing πριν από πέντε χρόνια, μου είπαν ότι είναι η πιο δύσκολη και σκληρή επιτροπή. Εκείνο που κατάλαβα στο πέρασμα του χρόνου είναι ότι αποτελείται από όλου εσά και του προκατόχου στην αίθουσα που διακρίνεστε για κοινωνική ευαισθησία και για ευρωπαϊσμό και σας ευχαριστώ για τη στήριξη της πολιτικής αυτής που έδωσε αποτελέσματα και θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από την καινούργια Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε. Actually, we have completed our timing. Πέρασε ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας για τη συνεδρίαση αυτή και υπάρχουν ακόμα κάποιοι ευρωβουλευτές που έχουν επιβιώσει και έχουν παραμείνει στην αίθουσα αυτή. Σας ζητώ συγγνώμη, χρειάστηκε να πάω στην Ολομέλεια για λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να εκφωνήσω ένα λόγο, επέστρεψα πάντως και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά, κύριε και κύριε Αβραμόπουλε. Επιτελέσατε το έργο σας, η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να είναι περήφανη που σας έχει και σας είχε επίτροπο για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι τόσο σημαντικό για μας, τόσο δύσκολο, τόσο ευαίσθητο Πραγματικά για πέντε χρόνια είχατε κεντρήσει την προσοχή μας και συμβάλλετε στο να μείνει όλη η συζήτηση ζωντανή. Θα θέλαμε λοιπόν να σας εκφράσουμε την θεσμική μας ικανοποίηση και δεν είναι απλώς, αν θέλετε, μία δείγμα ευγένεια μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά ειλικρινά θα θέλουμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την πολύ θετική συνεργασία που είχαμε και ελπίζω πραγματικά ότι θα υπάρξει και μια άλλη ζωή για σας, κύριε Αβραμόπουλε, μετά το τέλος της θητείας σας και θα θέλαμε πραγματικά να σας δούμε σε νέα αξιώματα, στα νέα αξιώματα που ενδεχομένω επιφυλάσσει για σας στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε. I'm, I'm